Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι η πρώτη συνεδρία της ομάδας μετά τις διακαπές, αλλά πριν από δύο ώρες, χάρη σε όλους σας, που είστε παρόντες εδώ ε, ήσασταν ε, σε συνδυασμένη ε, συνεδρίαση τριών επιτροπών για τη δασοκομεία και πριν αρχίσαμε με τις Space Policy διαπραγματεύσεις και μερικοί που ήταν συνάδελφοι εδώ εργάστηκαν. Εργαστήκαμε λοιπόν σκληρά σήμερα. Δεν έχουμε μόνο μέχρι το τέλος της θητείας τρεις συνεδριάσεις επιτροπής. Θα πρέπει να ε, το εκτιμήσετε αυτό πάρα πολύ. Ειδικό στις ψηφοφορίες. Καταλαβαίνω ότι το εκτιμάτε αυτό πάρα πολύ καλά και μερικοί από εμά που είμαστε από την Πολωνία είμαστε πολύ λυπημένοι απόψε το βράδυ αλλά θα πρέπει να υπερνικήσουμε τη λύπη μας και να προχωρήσουμε. Σας προτείνω λοιπόν να εργαστούμε σκληρά για να ενώσουμε την Ευρώπη μας. Ίσως το καταλαβαίνετε αυτό. Θα ήθελα να επανέλθω στη συζήτηση στην Ολομέλεια και σας ευχαριστώ πολύ που είστε παρόντες εδώ Όλοι πάρτε τις κάρτες σας, να τις βάλετε στη σχισμή, να δοκιμάστε τον τρόπο ψηφοφορίας. Χαίρεστε που είστε πάλι πίσω στο κοινοβούλιο μετά τις διακοπές. Ερώτηση που σας θέτω. Ναι, βεβαίως είναι ελεύθερη η ψηφοφορία εδώ. Αν αρχίζουμε την ψηφοφορία θα την αρχίζω και θα την κλείνω. Εντάξει. Α, Βλέπω είστε ευτυχείς. Θα ήθελα να πω ότι πρώτον θα υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη. Έχετε σχόλια. Δεν έχουμε σχόλια. Και περνάμε στο σημείο το 4, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρόκειται για την ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την ρομποτική. Εισηγητής ο συνάδελφος Ashley Fox και Περνάμε τώρα στην ε, διαδικασία ψηφοφορίας. Έχουμε συμβιβασμό α υπέρ, κατά αποχές ε, δεκτό. 49 υπέρ. Πρώτο τμήμα, πρώτο τμήμα, με συγχωρείτε. Υπέρ, κατά, αποχές, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Ας το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία και κλείνω την ψηφοφορία. Απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα. 50 υπέρ, κατά, αποχές. Ας το ελέγξουμε άλλη μια φορά. Άρχεται η ψηφοφορία και θα την κλείσω. Απορρίπτεται. F υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 55. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Ας το ελέγξουμε. Το πρώτο τμήμα. Κλείνω την ψηφοφορία. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, 59 ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 61 υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε. Συμβιβασμός 61. Καταπίπτει, καταπίπτει. Α, το 60 καταπίπτει, διότι αν το 51 γίνει δεκτός, το 60, ε, ο συμβασμός 60 καταπίπτει. 61. Κλείνω την ψηφοφορία. Δεκτή. G υπέρ, κατά, Αποχέσα. εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, ας το ελέγξουμε. Συμβιβασμός 76. Κλείνει η ψηφοφορία. 78 με τον 79 υπέρ κατά ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. Κλείνω την ψηφοφορία. 82 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό, 83, κατά, θα πρέπει, 83, 83 ελέγχουμε. Και κλείνει η ψηφοφορία. Συμφιβασμός δεκτός, 85 υπέρ, κατά αποχές γίνεται δεκτός H υπέρ κατά αποχές δεκτός J υπέρ κατά αποχές δεκτός ΕΝΚΟ 4 υπέρ κατά αποχές δεκτός ΕΝΚΟ 5 γίνεται δεκτός ΛΥΜΠΕ 14 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτός 95 υπέρ κατά αποχές δεκτός 96 πρώτο τμήμα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε 96 πέρα στις ψηφοφορίες Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. Ο 96. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. αποχέσα, Δεκτός. 101 υπέρ. Κατά. Δεκτό Δεκτός. Ε, των δύο υπέρ. Κατά. Δεκτός. Καίει. υπέρ. Κατά. Δεκτός. 114 υπέρ κατά αποχές δεκτός, 1.06 και κατά αποχές έγινε δεκτός, 1.17 υπέρ κατά αποχές δεκτός, συμβιβασμός L υπέρ κατά αποχές δεκτός, 125 υπέρ κατά αποχές δεκτός, M υπέρ κατά αποχές δεκτός, 129 υπέρ κατά αποχές δεκτός, 130 υπέρ κατά αποχές δεκτός, 132 υπέρ κατά δεκτός, 113 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτός. Γιούρι 3 υπέρ κατά αποχές δεκτός 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή 135 ε, δεκτή 139 ε, υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή 142 δεκτή 146 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 148 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 150 δεκτή ε, και πάλι δεκτή και έχουμε 140 κατά αποχές δεκτή, αποχές ναι, 144 δεκτή 145 υπέρ κατά αποχές δεκτή 149 υπέρ κατά αποχές δεκτή δεκτή 154 δεκτή ένα συμβιβασμός υπέρ κατά αποχές δεκτό Λίμπε 12 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά δεκτή ε, ο συμβιβασμός υπέρ κατά 166 υπέρ δεκτή 172 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 175 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 178 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ΙΜΚΟ 16 υπέρ ε, κατά ε, δεκτή, 153 υπέρ δεκτή, 179 δεκτή, ΙΜΚΟ 21, 182 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 183 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβασμός π και πάλι δεκτή, λίμπε 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 186 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 189 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 195 υπέρ, όχι, όχι, όχι, δεν ψηφίσαμε. 194 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 195 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 170 δεκτη 322 κατά αποχές δεκτή έχουμε συμβιβασμό Q υπέρ κατά αποχές δεκτή Γιούρι 4 υπέρ κατά δεκτή Γιούρι 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή MV4 υπέρ κατά δεκτή MV5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται MV6 υπέρ κατά αποχές, ας το ελέγξουμε. Και κλείνω την ψηφοφορία. MV9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, MV12 ε, κατά υπέρ κατά, α, θα πρέπει να ελέγξουμε για την MV12, MV12 και κλείνω την ψηφοφορία. Δεκτή, 200 υπέρ, κατά, δεκτή και πάλι δεκτή, 201 υπέρ, κατά, δεκτή, συμβιβασμός R υπέρ, κατά, δεκτή, 204 υπέρ, κατά, δεκτή, 205 υπέρ, κατά, α, ας ελέγξουμε. 205. Ελέγχουμε ε, και έκλεισε η ψηφοφορία 206 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ε, συμβιβασμός S υπέρ κατά δεκτός, 2, 1, 0 δεκτό, 2, 1, 1 υπέρ κατά δεκτή, 2, 1, 4 ε, υπέρ κατά δεκτή 2, 24, 2, 2, 3 υπέρ κατά δεκτή, 2, 2, 4 υπέρ κατά δεκτή. Περνάμε τώρα ε, στον συμβιβασμό τι υπέρ κατά Είμαστε σύμφωνα με το αλφάβητο στο τι. Λίμπε 17 υπέρ κατά αποχές 2-3-2 ε, υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε για την τροπολογία 2 2.32. Πώς ψηφίζουμε. Α, δεν σας βλέπω καλά. Πέρα της ψηφοφορίας. Α, λέτε σημαντικό, είναι σημαντικό. Α, απορρίπτεται, απορρίφθηκε. Δεν μπορώ να σας δω όλους βεβαίως. 2.34 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 2.35 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 2.43 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 2.44 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε. Γιατί 2.44. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται 2.45 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Φτάνουμε στο συμβιβασμό U υπέρ κατά αποχές δεκτός 2.47 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε 2.47 πέρα της ψηφοφορίας. απορρίφθηκε. 2.46 υπέρ κατά αποχέσα δεκτή. 2.60 υπέρ κατά δεκτή. Φτάνουμε στο, στο συμβιβασμό V στο W υπέρ κατά αποχές δεκτό, X υπέρ κατά αποχές δεκτός, Y υπέρ κατά αποχές δεκτός, Λίμπε 10 υπέρ κατά δεκτός 2.82 υπέρ κατά αποχές δεκτή Z ε, υπέρ κατά αποχές 2.87 ε, δεκτή ε, ΑΒ και πάλι δεκτή AC υπέρ κατά δεκτός AD υπέρ κατά αποχές δεκτός 3.1.1 Α, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ποιος το ανέφερε, ποιος ήταν τόσο γενναίος. Αγγερίτας. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Αλλά το λάθος μου, το λάθος μου κυρίως για σας. 304 ε, υπέρ κατά ε, δεκτή. AD υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3-1-1 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε. 3-1-1. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. 3-1-7 υπέρ κατά αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε για την 3-17. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. Φτάνουμε στο συμβιβασμό ΑΕ υπέρ κατά αποχές δεκτός, ΙΜΚΟ 3 ε, υπέρ κατά ΕΝΒ NV3 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε, 3-2-3 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 3-2-6 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 3.29 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 3.30 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ε, συμβιβασμός α δεκτή, εν, υπέρ, 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 11 υπέρ, θέλετε να ελέγξουμε, α 10, 10, ας ελέγξουμε γιατί 10. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. 11 υπέρ. Κατά δεκτή. 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ. Κατά αποχές. Α, δεκτή. 16 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 16 πέρα τη ψηφοφορία. Δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή, Συμβιβασμός Β υπέρ κατά αποχές δεκτός, 23 υπέρ δεκτός, 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 25 υπέρ κατά αποχές, ΙΜΚΟ Α υπέρ κατά αποχές δεκτή, ΙΜΚΟ Σ υπέρ κατά αποχές δεκτή, ΙΜΚΟ Δ υπέρ κατά αποχές δεκτή, ΙΜΚΟ Ε υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμχο F υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε. Γιατί νομίζω ίσως ο Πολ ψήφισε δύο φορές. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή ΙΜΚΟ G υπέρ κατά αποχές. Δεκτή MVB υπέρ κατά αποχές. Δεκτή MVC υπέρ κατά και πάλι αποχές απορρίπτεται MVD ε, ε υπέρ κατά αποχές δεκτή MVE υπέρ κατά αποχές δεκτή MVF υπέρ κατά θα πρέπει να ελέγξουμε MVF MVF και πέρα στις ψηφοφορίες Δεκτή, NVG υπέρ κατά αποχές η ίδια πλειοψηφία, αλλά στο ελέγξουμε άλλη μια φορά. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή MVH υπέρ κατά αποχές. Δεκτή MVI υπέρ κατά αποχές. Δεκτή MVJ υπέρ κατά ας ελέγξουμε. MVJ. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Συμβιβασμό C υπέρ, κατά αποχές δεκτός. 30 υπέρ κατά αποχές δεκτός, συμβιβασμός D υπέρ κατά αποχές δεκτός, 35 υπέρ κατά δεκτή, 36 υπέρ κατά δεκτή, 37 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε. 37. 37. Πέρα στις ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 41 υπέρ κατά δεκτή. 43 υπέρ κατά δεκτή. 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 5 υπέρ κατά ε, δεκτή, 6 υπέρ κατά δεκτή. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο ε, έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Πέραστης της ψηφοφορίας. Με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή. Αγαπητοί φίλοι, είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση για τις μελλοντικέ μας δραστηριότητες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τις μελλοντικέ δραστηριότητες της Επιτροπής μας στην επόμενη θητεία. Περνάμε τώρα στην απόφαση για την ενεργειακή απόδοση λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγητής είναι ο Μύροσλαβ Πόχε. Θα ψηφίσουμε unblock. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για την πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, όμως ε, είναι δυσάρεστο το παρελθόν της ε, έκθεσης και της ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια όμως Μύροσλαβ. Ψηφίζουμε τώρα για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων. Άρθρο C, επίση με ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Ξέρετε πως ιδιαίτερα για μένα είναι αρκετά λυπηρό το ιστορικό της ψηφοφορία αυτής. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ τον Μύροσλαβ. Περνάμε στον Ενίσα πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η συγκήτρια Εγγέλικα Νίμπλερ είναι μαζί μας και ψηφίζουμε την προσωρινή συμφωνία στην οποία οδηγήθηκε ο τριμερής διάλογος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Εξαιρετικό αποτέλεσμα όπως και όλα τα προηγούμενα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Αγγέλικα και σε όσους συμμετείχαν στην πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Φρέντερικ Φέντερλεϊ, υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επίπεδου.eu. Ψηφίζουμε για την προσωρινή συμφωνία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Συγχαρητήρια, Φρέντερικ. Εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αγαπητοί φίλοι, εκτιμήσατε λοιπόν αυτή την ψηφοφορία, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί δεν μας μένουν πολλές μέχρι τη λήξη της θητείας, είναι μία από τις τελευταίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε όμως και τη συνέχεια της ε, συνεδρίασης τη επιτροπή μας. Ένα ακόμα σημείο στην ημερησία διάταξη. Είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι. Απίστευτο. Θα σας παρακαλούσε, λοιπόν να απομακρυνθείτε αθόρυβα. Αν θέλετε φυσικά να απομακρυνθείτε και να εξαφανιστείτε, διότι θα προτιμούσα να μείνετε όλοι εδώ μαζί μας. Okay, okay, let us start. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σύσταση του... Πόπο. Δεν γίνεται, δεν γίνεται να προχωρήσουμε. Point 8. Σημείο 8. Στην ημερήσια διάταξη. Σύσταση του Ευρωπαϊκού Βιομηχανικού, Τεχνολογικού και Ερευνητικού Κέντρου Ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνασφάλειας και του δικτύου Εθνικών Κέντρων Συντονισμού. Η συγγήτρια είναι η Γιούλια Ρέντα. Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ε, περσινό Σεπτέμβριο του 2018 και συνδέεται με το ε, απερχόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρόκειται για την δημιουργία ενός ε, οργανισμού για την ε, ασφάλεια, αλλά και για τα το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη. Είναι δύο προγράμματα για τα οποία είναι αρμόδια η Επιτροπή μας. Δεν θα σταθεί δυνατό να ολοκληρωθούν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις πριν το τέλος της ε, κοινοβουλευτικής θητείας, όμως ε, θα καταφέρουμε, ελπίζω, να ολοκληρώσουμε την, ε, το δικό μας μέρος μέχρι τον Απρίλιο για να διευκολύνουμε τη δουλειά του επόμενου Ευρωκοινοβουλίου. Όπως γνωρίζετε, η κυβερνασφάλεια είναι ιδιαίτερα σημαντική και η συγκήτρια έχει 113 τροπολογίες στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε στη διάθεσή μας μισή ώρα περίπου για την συζήτηση, όμως δεν θα πρέπει να τελειώσουμε μετά τις 10 και μισή. Έχετε μία ώρα αν θέλετε να το συζητήσετε. Κύριε Ρέντα, λοιπόν, θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους που αποφάσισαν να μείνουν αυτή την περασμένη ώρα για την συζήτηση του θέματος αυτού. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μην εξαντλήσω ότι είναι μία ώρα που μας μένει, να μην συζητήσουμε και τις 113 τροπολογίες. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Βιομηχανικού, Τεχνολογικού και Ερευνητικού Κέντρου Ικανοτήτων στον τομέα τη κυβερνοασφάλεια και του Δικτύου Εθνικών Κέντρων Συντονισμού. Από εδώ και στο εξή θα ε, αναφέρεται ω CCEN. Αφορά υποδομές και υπηρεσίες που έχουν σχέση με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Όλο ένα και περισσότεροι καταναλωτές συμμετέχουν στο διαδίκτυο των πραγμάτων και αυτό λοιπόν ε, έχει αλλάξει τα δεδομένα. Το 2016 ξεκίνησε μία ε, νέα, η χρήση μιας νέας ε, τεχνολογίας που πολλοί από εμά την έχουμε ήδη στα σπίτια μας. VPN είναι πολύ σημαντική για την επικοινωνία, την συμμετοχή μας στα ε, στο κοινο... στην κοινωνία. Είναι βασισμένη λοιπόν σε ορισμένα βασικά συστατικά στοιχεία που βρίσκονται σε διαφορετικά προϊόντα. Πολλά από αυτά τα συστατικά στοιχεία μέχρι και τις εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιούμε δημιουργούνται από κοινότητες ε, ανοιχτού λογισμικού. Υπάρχουν ευάλωτα λοιπόν ε, σημεία στη χρήση αυτού του ανοιχτού λογισμικού, όμως η τεχνολογία μπορεί να μας φτάσει πάρα πολύ μακριά. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω το κέντρο αυτό να αυξήσει την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια του ε, υλικού και του λογισμικού, ιδιαίτερα του ελεύθερου λογισμικού και υλικού για την αύξηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Η πρόταση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πώς ε, θα δημιουργηθεί το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εκείνες ε, που αναπτύσσουν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό το λογισμικό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, όμως δεν είναι οι μόνες. Υπάρχουν και πάρα πολλές ε, μεγάλες επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις γεμάτες καινοτομία. Πολύ συχνά, επίσης, η πανεπιστημιακή κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών δίνουν το ένασμα για περαιτέρω έρευνα. Χρειάζεται λοιπόν να αναγνωρίσουμε αυτήν την συμβολή της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς επίσης και το ότι οι απειλές στον κυβερνοχώρο είναι υπαρκτό φαινόμενο που απειλούν τους ε, πολίτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο, δεν μπορούμε να αποδώσουμε με βεβαιότητα μία κυβερνοεπίθεση σε μια συγκεκριμένη οντότητα. Οι κυβερνοεπιθέσεις πολλές φορές μας οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα σχετικά με την προέλευσή τους. Γι' αυτό το ΝΑΤΟ και άλλοι οργανισμοί εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήση συμβατικών μεθόδων για την αντιμετώπιση των απειλών αυτών. Υπάρχουν, είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη αμυντικούς σκοπούς να μην ε, χορηγείται σε ε, έρευνα που σχετίζεται και με θέματα άμυνας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Επίσης, αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρώπη να προάγει τα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ε, τις αξίες της και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να αυξηθεί η και η ακεραιότητα των συστημάτων, ενώ από την άλλη επιθετικά στρατιωτικά προγράμματα είναι κάτι το οποίο είναι αντίθετο προς τον σκοπό αυτών. Και σε πολιτικό και σε στρατιωτικό πλαίσιο υπάρχουν ορισμένα προϊόντα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και αυτά χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες ε, επικοινωνίας και πληροφορίας. Επίσης, χρειαζόμαστε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη καθώς και μεγάλες ανισορροπίες ως προς την ε, εκπροσώπηση των ε, φύλων αλλά και την γεωγραφική κατανομή των εργαζομένων. Τέλος, την έκθεσή μου ζητώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ίση θέση με τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την λήψη αποφάσεων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε μόλις το Σεπτέμβριο, γι' αυτό δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί το θέμα με τριμερείς διαλόγους πριν τις ευρωεκλογέ. Από όσο γνωρίζουμε, το Συμβούλιο θα εξετάσει το θέμα από το Μάρτιο, όμως ε, δεν θα φτάσει ο χρόνος για να μπούμε σε τριμερεί διαλόγου μέχρι τις ευρωεκλογέ. Γι' αυτό ελπίζουμε να υιοθετήσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία θέση μέχρι τις ευρωεκλογέ έτσι ώστε το θέμα να προχωρήσει από τον Ιούλιο. 16 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες. Και φυσικά για να επιτύχουμε το στόχο αυτό πρέπει όλοι να συνεργαστούμε άριστα. Ελπίζουμε λοιπόν το Μάρτιο να εγκρίνουμε στην πρώτη ανάγνωση το ε, θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, παρουσίαση της έκθεσής σας. Πάμε τώρα στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων από το ΕΛΚ. Ο Πολ Ρούμπικ. Έχασε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εισηγήτρια, διότι πιστεύω πως είναι επίγουσα ανάγκη να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Έχουμε δει ότι μπορούν να προκληθούν σοβαρές ζημιές από απειλές στον κυβερνοχώρο. Για τον λόγο αυτό, έχουμε εξετάσει το θέμα από πολλές οπτικές γωνίες. Υπάρχουν τέσσερις μελέτες ε, οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα αυτό και νομίζω πως αποτελούν μια πάρα πολύ καλή βάση η πρώτη έχει να κάνει με την ε, αυτόματη αντιμετώπιση παρά της παραπληροφόρησης. Ασχολείται με ζητήματα ποιότητας, ποσότητας, με τις επιπτώσεις ε, της χρήσης αλγορίθμων, ε, οι οποίοι διανέμουν πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, να δούμε σε επίπεδο πολιτικής και δημοκρατίας ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός ε, εάν, ε, ανάμεσα σε στρατιωτικό και πολιτικό σκέλος. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό η αυτοματοποίηση να σταθεί στο επίκεντρο του ε, ενδιαφέροντός μας. Έπειτα, δεύτερη μελέτη, αλγόριθμοι, προκλήσεις και ευκαιρίες. Η μελέτη αυτή ασχολείται με τη διαφάνεια και την ιεράρχηση των ε, αλγοριθμών, οι οποίοι στο μέλλον θα παίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η μελέτη λοιπόν αυτή δείχνει ξεκάθαρα, πιστεύω, ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε, αλλά και ποιες είναι οι προκλήσεις. Μετά, η επόμενη μελέτη, πλαίσιο διακυβέρνησης για τους ε, αλγόριθμους και την αύξηση της διαφάνειας. Δηλαδή, τι μπορούμε να ρυθμίσουμε ε, σε τεχνικό επίπεδο, ποια είναι τα σημαντικά θέματα που μπορούν να λυθούν, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ε, ποια μέτρα θα μπορούσαν να έχουν εθελοντικό χαρακτήρα. Τι μπορεί να κάνει η πολιτική λοιπόν, να εξετάσει, κατά την άποψή μου, τους ε, τομείς και να αποφασίσει για το που χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση και που όχι. Επίσης, υπάρχει η τελευταία μελέτη για την ε, πολιτική άμυνας και την ε, άμυνα στον κυβερνοχώρο. Η μελέτη αυτή δείχνει τις ε, δυνατότητες και στον στρατιωτικό άξονα και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η έρευνα και η επιστήμη. Επίσης ασχολείται με την αύξηση της διαφάνειας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Η τελευταία λοιπόν μελέτη έχει να κάνει με την ε, νομοθεσία, παραπληροφόρηση και τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω πως αυτή η μελέτη είναι μια πάρα πολύ καλή προσθήκη στην έκθεση πρωτοβουλίας μας, διότι φυσικά προσπαθούμε και τα 28 κράτη-μέλη να συνεργαστούμε έτσι ώστε να αποφύγουμε την φοροδιαφυγή και την φόρο αποφυγή. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμός ε, μεταξύ των 28 κρατών μελών. Εδώ δημιουργούνται προβληματισμοί σχετικά με την δομή που θα πρέπει να έχει ένας τέτοιος οργανισμός. Υπάρχουν προτάσεις για διάφορα μοντέλα ε, και για διάφορα στάδια. Σε πρώτο στάδιο πιστεύω θα πρέπει να αποφασιστεί η αρχιτεκτονική του υλικού και του λογισμικού, να γίνουν καλυστία ε, εντό εισαγωγικών των βέλτιστων πρακτικών, έτσι ώστε να κερδίσει ο καλύτερος. Έπειτα, δεύτερο στάδιο, παραγωγή, εγκατάσταση του λογισμικού, εγκατάσταση του υλικού. Αυτό πρέπει να γίνει από ανεξάρτητες εταιρείες και σε τρίτο στάδιο συντήρηση και χρήση των συστημάτων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν μετά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση να διασφαλίζεται και η σωστή ε, συντήρηση και σωστός έλεγχος. Χρειάζεται λοιπόν αντικειμενικότητα ως προς τον έλεγχο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και πιστεύω πως θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό εκτός από την ε, πολιτική να συμμετέχει στον έλεγχο και ε, ένας εκπρόσωπος των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται αυτή η διαφάνεια. Έτσι νομίζω θα καταφέρουμε, συνδυάζοντας όλα αυτά, να συντάξουμε μία μελλοντοστραφή έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σου και τις συγκεκριμένες προτάσεις σου και τα αποτελέσματα της έρευνας που μας παρουσίασε. Πολλά είπες. Αυτό τι σημαίνει όμως ότι και όλοι οι υπόλοιποι έχουν απεριόριστο χρόνο. Ισότητα. Ίδιες δυνατότητες λόγου, έτσι. Απεριόριστος χρόνος για όλους και για την εισηγήτρια. Ποιος είναι ο επόμενος? Ο επόμενο, κυρία Γκρίφιν, από του σοσιαλιστέ. Απεριόριστο χρόνο. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ δημοφιλή αν ε, χρησιμοποιήσω απεριόριστο χρόνο. Τέλο πάντων, ε, ο σκιώδη εισηγητή μα, ε, Γιάνν Γκάιερ, δεν μπόρεσε να έρθει εδώ. Είναι στο Βερολίνο και τον εκπροσωπώ. Πριν όμω, Γέρζη, ξεκινήσω την ομιλία μου εξ ονοματό του να σα συλληπιθώ για τα τραγικά συμβάντα στην Πολωνία τις τελευταίε δύο μέρε. Και για το Brexit, φυσικά θα το σχολιάσω το θέμα. Είναι θλιβερό που πρέπει να ψηφίσουμε για να προσαρμόσουμε την ε, οδηγία ε, λόγω της αποχώρησης του Brexit, αλλά υπάρχει ελπίδα. Ε, μπορεί και τον Ιούλιο να είμαστε ακόμα εδώ. Ελπίζω. Φυσικά, εμείς οι σοσιαλιστές θα θέλαμε να είμαστε ακόμα τμήμα της θαυμάσιας αυτής κοινότητας. ορίσουμε την πρόταση να δημιουργήσουμε, δημιουργήσουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βιομηχανικού, Τεχνολογικού και Ερευνητικού ε, ερευνητικών ικανοτήτων ε, είναι σημαντικό για την Ευρώπη, ε, για την ηγεσία της Ευρώπης, ούτως ώστε να προστατεύσουμε τους πολίτες και την οικονομία μας αποτελεσματικά εναντίον των ε, όλων και αυξανόμενων κυβερνοεπιθέσεων. Πιστεύουμε ότι το κέντρο ικανοτήτων μαζί με το, την κοινότητα ικανοτήτων και τα εθνικά κέντρα συντονισμού είναι ένα βασικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Ρέντα για την έκθεσή της. Ε, συμφωνούμε πολλές από τις ιδέες της ε, και κάποιες από τις οπολογίες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Φερρυπίνη ό,τι αφορά μια πιο ολιστική προσέγγιση για την ε, κυβερνοασφάλεια και την προστασία των πολιτών αυξάνοντας την αφύπνιση, την εκπαίδευση ε, και να δώσουμε και περισσότερο λόγο ε, στο Κοινοβούλιο για το Κέντρο Ικανοτήτων. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν και κάποιες προσαρμογές που θα πρέπει να γίνουν στην πρόταση της Κομισιόν. Υποστηρίζουμε ε, τις έξι ενέργειες μεταξύ ε, των λύσεων της κυβερνοασφάλειας ε, στον τομέα της άμυνας και το μη αμυντικό τομέα. Πιστεύουμε όμως ότι είναι σημαντικό να εγγυηθούμε ότι η ψηφιακή Ευρώπη και ο ορίζοντας Ευρώπη χρησιμοποιούνται μόνο για μη στρατιωτικά έργα. Θα πρέπει λοιπόν τα έργα διτής χρήσεως να χρηματοδοτούνται από το αμυντικό ταμείο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εκεί τις προτεραιότητες μας για την άμυνα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται ε, να είναι στο κέντρο της προσοχής του κέντρου, ε, γιατί είναι βασική εταίροι ε, για την κυβερνοασφάλεια και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια, συνοχή με άλλες ευρωπαϊκές δράσεις για την κυβερνοασφάλεια και με άλλους φορείς όπως τον ΕΝΙΣΑ και θέλουμε και οι υπάρχουσες δομές όπως η ΕΞΚΟ να παίξουν σημαντικότερο ρόλο στο κέντρο και, στο, και στην κοινότητα ικανοτήτων γιατί πιστεύουμε ότι δεν έχουν ε, εξεταστεί σωστά από την Κομισιόν μέχρι στιγμής. Ένα άλλο σημείο είναι ότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή ηγεσία. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να περιορίσουμε την ε, συμμετοχή στο κέντρο σε εταιρείε ε, με έδρα στην Ευρώπη ή στον ΕΟΧ ή στην ΕΖΕΣ και ελπίζουμε και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίση, ε, συμβουλευτικό ρόλο θα πρέπει να έχει ο κλάδο ε, και τα συνδικάτα γιατί έχουν πυρογνωμοσύνη στον τομέα. Προσβλέπουμε σε συνεργασία με τον εισηγητή, με την εισηγήτρια και με του κοιόδη εισηγητέ για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Τερέζα, για την ε, παρουσίασή σου εξ ονόματος του συναδέλφου. Τώρα περνάμε στην ε, ομάδα μεταρρυθμιστών και συνδυστών ο συνάδελφος Σουσανόφσκι που αντικαθιστά κάποιον. Ναι, σας δίνω λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα <clears throat> να ευχαριστήσω την εισηγήτρια η οποία προχώρησε αρκετά το θέμα. Θα ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα τα οποία είναι ερωτηματικά για μένα. Η κυρία Ρέντα ε, ε, εστιάζεται ε, πιο πολύ στην χρήση την πολιτική και όχι τη στρατιωτική. Το συζητήσαμε αυτό στο παρελθόν, αλλά ο χρόνος μας δείχνει ότι ορισμένες αλλαγές είναι απαραίτητες και Έχουμε βεβαίως την κυβερνοασφάλεια, την κυβερνοάμυνα που απαιτούν κάποιο σχέση, κάποιο σύνδεσμο με τα αμυντικά συστήματα, κάποια συνδεσιμότητα με τα ε, συστήματα αυτά ε, πολιτικά και αμυντικά, στρατιωτικά που δεν μπορούν να διαχωριστούν διότι η κυβερνοασφάλεια και η κυβερνοάμυνα πρέπει να περιλαμβάνουν ε, σύνδεση με τον στρατιωτικό τομέα και με τον πολιτικό. Αυτά όλα είναι συνδεδεμένα. Δεν νομίζω ότι ε, θα πρέπει να έχουμε πέντε μέλη στο Συμβούλιο. Έχουμε ασχοληθεί ε, με το θέμα σε σχέση με άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες και δεν νομίζω ότι το Κοινοβούλιο χρειάζεται ε, να είναι εδώ στο Συμβούλιο, διότι χρειάζεται μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη ε, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει η Κομισιόν να έχει 50% των ψήφων, διότι αυτό θα δώσει ένα δικαίωμα βέτο στην Κομισιόν. Πιστεύω ότι η αντιπροσώπευση των κρατών μελών ανάλογα με την οικονομική του συνεισφορά δεν είναι νομίζω και αυτό μια καλή λύση. Ενίσα, ο Ενίσα γίνεται ένα είδος κέντρου, κέντρου για ολόκληρη την Ευρώπη. Και νομίζω, πιστεύω, ότι περισσότερο άνοιγμα, περισσότερο συντονισμός με φιλικές τρίτες χώρες θα ήταν μια καλή λύση. Ίσως θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί. Ευχαριστώ την κυρία Ρέντα που μπόρεσε να προχωρήσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αγγέλικα Μίλνερ ε, έχει την ευθύνη για την ομάδα Άλτα. Ευχαριστώ. Δεν θα έχω μια ανοιχτή προσέγγιση. Θα προσπαθήσω να είμαι ε, σύντομη και συνοπτική. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης και για τα σχόλια των συναδέλφων. Έχουμε όλοι έτσι κάπως μια εντύπωση για τον προσανατολισμό των διαφόρων ομάδων. Ε, χαιρετίζω το σχέδιο έκθεσης σε σχέση με τον ρόλο που αποδίδεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στη διακυβέρνηση και μεγαλύτερη συνέπεια των προτάσεων σε σχέση με το πλαίσιο πολιτικής εξασφαλίζοντας την ε, συμπερίληψη του ΕΝΗΣΑ σε ε, σχέση ε, με τις πρόσφατες εξελίξεις της, του οργανισμού. Επίσης, καλή αντιπροσώπευση όλων των πρωταγωνιστών της κοινότητας κυβερνοασφάλειας. Δύο συνάδελφοι είπαν ότι θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω τον περιορισμό ίσως της εφαρμογές του πολιτικού τομέα. Σύμφωνα με την ομάδα μου αυτό ίσως θα μπορούσε να έβλαπτε την πρωτοβουλία αυτή καθε να και ίσως αποκλείεται έτσι η χρηματοδότηση από άλλες πηγές, διότι έχουμε και εφαρμογές βιομηχανικές και στρατιωτικές και θα χάσουμε και την εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει στον τομέα των δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας ως ηγήτρια ε, για τα δύο δισεκατομμύρια που έχουμε για την κυβερνοασφάλεια που θα χειρίζεται το κέντρο κυβερνοασφάλειας. Ελπίζω ότι θα υπάρξει συντονισμός ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο, τα Εθνικά Κέντρα Συντονισμού ε, και το Κέντρο Digit Innovation ε, που θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα το ψηφιακό. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε μια προσπάθεια για να υπάρξει κάποια συνέργεια ανάμεσα σε αυτούς που θα μπορούν να ωφεληθούν από όλα αυτά. Αυτό είναι έργο μας, καθήκον μας να τα εξασφαλίσουμε όλα αυτά. Περιμένω με ενδιαφέρον την, συνεργασία με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Ο Αντιπρόεδρος, κύριος Κοχίτσε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Πολύ ωραία, θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, τα τσέχικα. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε ο κ. Κοσενόφσκι και Μινάρ. Έχουν πρόβλημα με την ε, διπτή χρήση της τεχνολογίας. Η τσεχική δημοκρατία είναι έδρα μία από τις μεγαλύτερες ε, υπηρεσίες ή οργανισμούς κυβερνοασφάλειας. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν η εκπροσώπηση αυτή να μην βασίζεται στο μέγεθος της συνεισφοράς, δηλαδή της γραμμής του προϋπολογισμού, αλλά να υπάρχει ίση εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών, μια και όλα τα κρατημέλη έχουν ίσα δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά αυτά που είπε η Βρετανίδα συνάδελφος, η συνεργασία πιστεύω ότι θα συνεχιστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, η κυβερνοασφάλεια είναι ένα παγκόσμιο μέλημα, δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ηνωμένο ή τη Ρωσία, τις Ηνωμένε Πολιτείε ή την Ιαπωνία. Είναι ένα παγκόσμιο θέμα το οποίο θα πρέπει να μα απασχολήσει όλους από κοινού, ανεξάρτητα της ιδεολογίας μας. Είναι θέμα ασφάλεια όλων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γερομίλ, για τα όσα είπες. Η Αυστριακή αντιπροσωπεία, όσα και η Κυρία Κάπελ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, πράγματι φαίνεται πως η Αυστρία έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ε, κυβερνοασφάλεια. Αυτό φάνηκε κιόλα. Ε, πάντως, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και όλους τους εισηγητέ. εισηγητές. Ε, νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να εργαστούμε πάνω στο φάκελο αυτό ε, πριν τη λήξη αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε οι ικανότητες να παραμείνουν εντός Ευρώπης στον ε, τομέα αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται και ένα κέντρο ικανοτήτων ε, αντί για πολλά εθνικά κέντρα. Αυτό το κέντρο λοιπόν θα πρέπει να λειτουργήσει ως κολαπτήριο ιδεών και ε, προτάσεων νέων φρέσκων προτάσεων για την βελτίωση της κυβερνοασφάλειας. Βλέπουμε πως η απειλές ναι. ένα και αυξάνονται. Υπάρχουν ε, μικρότερες και μεγαλύτερες επιθέσεις, ε, κυβερνοεπιθέσεις και αυτό δείχνει πως χρειαζόμαστε αύξηση των ικανοτήτων μας στην ε, άμυνα στον χώρο. Χρειάζεται λοιπόν να χαράξουμε νέους δρόμους και το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να αποτελέσει τον κόμβο και το κέντρο αριστείας υπό τον ε, ορίζοντα Ευρώπη. Νομίζω πως ε, φαίνεται η σημασία της δημιουργίας ενός τέτοιου κέντρου. Ήδη αναφέρθηκαν από πολλούς ε, συναδέλφους πολλά τα οποία ήθελα να αναφέρω κι εγώ. Ενίσα, για παράδειγμα, εδώ πρέπει να τονίσω πως δεν έχουν δεν έχουμε σκοπό να ε, πάρουμε αρμοδιότητες από τον ΕΝΗΣΑ, αλλά να λειτουργούν αυτοί οι δύο οργανισμοί συμπληρωματικά. Χρειάζεται επίσης να προσέξουμε να μην χαθεί χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα, καθώς και να μην χαθεί εμπειρογνωμοσύνη. Η διτή χρήση είναι πολύ σημαντική και δεν πρέπει να την προσπεράσουμε όταν μιλάμε για κυβερνοασφάλεια. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι κάτι το οποίο ήθελα να δεν νομίζω πως χρειάζεται απαραίτητα πέντε μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε και πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει το ίδιο δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα βέτο με τα κρατη Αυτά λοιπόν τα τρία σημεία νομίζω είναι τα σημαντικότερα. Αναφέρθηκαν και από αρκετούς. Ε, ελπίζω οι εισηγήτρια και οι εισηγητές να καταλήξουν σε μια πολύ επικοδομητική έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Δεν θέλει κάποιος ε, το λόγο, από την Αυστρία τουλάχιστον, άρα κανείς μάλλον. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο Γκοντζάλε Σάντσο από την ε, DigiConnect. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Ρέντα για την έκθεσή σας. Ευχαριστώ όλους όσους μίλησαν υποστηρικτικά υπέρ της πρότασης Κομισιόν. Σημείωσα κάποια σχόλια στα οποία θα ήθελα να σταθώ για το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Φερρυπίν, που τονίσατε πολύ από εσά. Συμφωνώ και συμφωνεί αυτό που είπατε με το πνεύμα και το γράμμα της ε, πρότασης. Στην έκθεση Ρέντα δίδεται σημασία στην ε, σημασία ανοιχτού λογισμικού, ελεύθερου λογισμικού ανοιχτής πηγής. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει το θέμα της εκπροσώπησης, της αντιπροσωπευτικότητας που αναφέρατε πολύ από εσά. Αυτό θέλει και η Κομισιόν. Αντιπροσωπευτικότητα. Το θέμα είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία, απλώ. Να υπάρχει ευρύ εκπροσώπηση, αλλά και να έχουμε και δομέ οι οποίε θα λειτουργούν. Αυτό που είναι σημαντικό, να υπάρχει και η κατάλληλη πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα εκπροσωπείται στις δομές. Θα πρέπει να βρούμε αυτή την ε, αντιπροσωπευτικότητα, λοιπόν. Φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει λόγο και να εμπλακεί στο σύστημα για το θέμα της άμυνας και τις σχέσεις με τα αμυντικά. Αυτό είναι μια δομή μη στρατιωτικού χαρακτήρα για να υπάρξει χρηματοδότηση. Και οι κανόνες που θα ακολουθηθούν θα είναι αυτοί των προγραμμάτων χρηματοδότησης του ορίζοντα δηλαδή 2020 και, του, και της ψυχιακής Ευρώπης. Υπάρχει δυνατότητα όμως και άλλα προγράμματα να συμβάλλουν για την συμπληρωματικότητα με την ΕΝΗΣΑ. Φυσικά, η ΕΝΗΣΑ είναι τμήμα του όλου συστήματος. Αναφέρατε το ρόλο ε, της Κομισιόν και το δικαίωμα ψήφου που έχει η Κομισιόν. Σε αυτή την πρόταση έχουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και επιπλέον χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν παρετείται από το δικαίωμα πρωτοβουλίας τροποντινά σε αυτό το κέντρο. Όμως ε, εμείς είμαστε ο θεματοφύλακας των, του ενωσιακού προπολογισμού. Και ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε κάποιο λόγο. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι για τις δυσκολίες των διαπραγματεύσεων σε, σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Είναι πρόκληση αυτό, είναι δύσκολο, αλλά συνεργαζόμαστε και με το Συμβούλιο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πέρα ή δυνατόν από την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο με το Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν φυσικά ε, προτίθεται να κάνει ό,τι μπορεί για να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις αμελητή. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Την ίδια πρόθεση έχουμε προφανώς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τζούλια, απεριόριστο χρόνο στη διάθεσή σου έχεις. Ε, κάποια στιγμή θα φεύγει και ο κόσμο. Ε. Θέλω να ευχαριστήσω του Σκιώδη για τι επικοδομητικέ παρατηρήσει του. Πολλά σημεία σύγκληση έχουμε. Συμφωνούμε να υποστηρίξουμε αυτή τη νέα δομή, εξασφαλίζοντα ότι δεν θα κανιβαλίσει τι λειτουργίε του ΕΝΗΣΑ, που είναι πολύ επιχειρησιακό οργανισμό. Εδώ μιλάμε για την χρηματοδότηση και την κατανομή τη χρηματοδότηση περισσότερο. Υπάρχουν κάποια δύσκολα ερωτήματα για την άμυνα και τη σχέση ανάμεσα στους διάφορους προϋπολογισμούς. Συμφωνούμε όλοι φυσικά ότι θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες για το, την ψηφιακή Ευρώπη και τα προγράμματα ορίζοντας Ευρώπη που δεν θα πρέπει να ξοδεύουν τα λεφτά τους για την άμυνα. Συμφωνώ ότι οι τεχνολογίες διπλής χρήσης είναι αναπόφευκτες. Δεν θα πρέπει να μπουν σε αυτή την πρόταση, όμως είναι η χρηματοδότηση για επιθετικές τεχνολογίες. Ε, που υποσκάπτουν την ασφάλεια παρά την ενισχύουν. Και επίσης είμαι λίγο διστακτική για τις υποχρεώσεις της συνθήκη και για το κατά πόσο μπορούν να γίνουν σεβαστέ. Εάν φτιάξουμε μια δομή ότι η χρηματοδότηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμυνα, αλλά η δομή αυτή θα μπορεί να διαχειρίζεται ε, κονδύλια τα οποία έχουν ε, ήδη εκ των προτέρων προοριστεί για την άμυνα. Κοιτάω λοιπόν λίγο του σοσιαλιστές για να δω πώς θα μπορέσουμε από κοινού να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις υποχρεώσεις τη συνθήκη ε, της συνθήκης, ώστε τα λεφτά τα οποία προορίζονται για μη στρατιωτικού σκοπούς να ξοδεύονται για μη στρατιωτικού σκοπούς. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ όλους 16 Ιανουαρίου 2019, 12 η ώρα, είναι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες. Επόμενη συνεδρίαση θα είναι 23 Ιανουαρίου και 24 θα ίσως ε, θα περιοριστεί ή ίσως και θα καταργηθεί αυτή η συνεδρίαση, αλλά 23 Ιανουαρίου θα έχουμε ασφαλώς ε, μία συνεδρίαση της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ωραία. Ελπίζω να υπάρχει. Ναι, καλά ήταν και αυτό το λιγότερο.